Good morning. Καλημέρα σας. Άρχεται η συνεδρίαση. Έγκριση μερίσια διάταξη είναι το πρώτο θέμα. Εάν δεν επιθυμείτε αλλαγέ, εγκρίνεται όσο έχει ημερήσια διάταξη. Το δεύτερο σημείο. Ανακοινώσει της Προέδρου και συστάσει των συντονιστών στις 25 Απριλίου οι ε, συντονιστές αποφάσισαν να συντάξουμε έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για την εσωμάτωση ε, του φίλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με εισηγήτρια την κυρία Μιλίναρ από τους φιλελευθέρους. Επίσης για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, άλλη έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας ε, 2016-2017 να δοθεί στους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ε, νομοθετική γνωμοδότηση για την έκθεση της Επιτροπής ΕΜΠΕΛ ε, για την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Αρχής ε, Απασχόλησης και να πάρουν αυτό το θέμα οι πράσινοι. Επίσης εκπώνηση μάλλον τροπολογιών στην νομοθετική έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας των αστυνομικών ταυτοτήτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αδειών ε, παραμονής σε εκείνους που διαμένουν σε άλλη χώρα από την πατρίδα τους και να την αναλάβει αυτή η ε, ομάδα των φιλελευθέρων. Επίσης, γνωμοδότηση στην ε, έκθεση της πρωτοβουλίας ΑΦΕΤ για την εποχή μετά την Αραβική Άνοιξη στη Μέση Ανατολή για τον πάνω σοσιαλιστές και δημοκράτες έκθεση δίας πρωτοβουλίας της Επιτροπής ΕΚΟΝ να κάνουμε γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την ετήσια ανάπτυξη ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Προφορική ερώτηση με ψήφισμα για την οπισθοδρόμηση στα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΓΚΟΕ. Προφορική ερώτηση με ψήφισμα για την κατάσταση και τα δικαιώματα των γυναικών με αναπηρίες το ΕΛΚ. Και μετά από σύγκρουση αρμοδιοτήτων με την Επιτροπή Απασχόληση, ο τίτλο τη ε, έκθεση ιδέα πρωτοβουλία μα για ε, την ε, ισορροπία εργασιακού και ιδιωτικού βίου έχει αλλάξει. Επόμενο θέμα, η έγκριση των πρακτικών 19 και 20 Φεβρουαρίου και 8 Μάρτιου. Εάν δεν έχετε άλλα σχόλια, θεωρούνται τα πρακτικά εγκεκριμένα. And Τέσσερα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι να ψηφίσετε συνάδελφοι. Παρακαλώ, ετοιμαστείτε για να αρχίσουμε αμέσω να ψηφίζουμε. Okay. Yeah. Uh... Σημείο 4. Η κατάσταση στην Ουγγαρία. Σε συνέχεια του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη 17 7η Μαΐου 2017. Η τροπολογία 29. Ψηφί υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. Η τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 47 με μια προφορική τροπολογία της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Τροπολογία 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά απόχες εγκρίνεται. Η συμβαστική 7 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 65 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπάρχει 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 ε, με προφορική τροπολογία της ηγήτρας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 93 και 94 ταυτίζονται υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 3 με προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 4 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 6 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 8 είπε, κατά αποχές έλεγχος χρειάζεται εδώ. Αρχίζει τώρα. And now the vote is Πέρας. It's adopted. Ε, Η τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 11 υπέρ. Against abstention. Ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 21 σε διατμήματα, τμήμα πρώτον υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και οι 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία τελική για το σύνολο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει τώρα. And now the vote is... Εγκρίνεται η γνωμοδότηση χαρητήρια κυρία Νόιχελ και σκιώδης συγγητέ. σα ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο σημείο 5. Συνοπτική έκθεση των προτεραιοτήτων της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των φίλων. Πρώτη παράγραφος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη παράγραφος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5 Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12, εδώ έχουμε προφορική τροπολογία, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ.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 Περνάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές. Εδώ συντάκτρια γνωμοδότησης είναι η Ανιέσκα Κρουσλόφσκα Θα εξετάσουμε εδώ πέρα τις τροπολογίες. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Κοσλόφσκα Ραγεβίτς. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό σχέδιο γνωμοδότησης. Ελπίζω ότι ε, η άδεια πατρότητας και η γονική άδεια θα ισχύουν παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κατάλληλες αμοιβέ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές, όλους τους συνεισηγητές και όλους όσοι συμμετείχαν στη σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης. Υπήρχαν πολλοί συνάδελφοι από την Επιτροπή μας που συμμετείχαν στην όλη διαδικασία και αυτό φαίνεται και από τις πάρα πολλές τροπολογίες που κατατέθηκαν. Η Επιτροπή Απασχόλησης είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή για την έκθεση αυτή. Η δική μας η Επιτροπή από την άλλη είναι υπεύθυνη για την σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης. 473 συνολικά είναι που κατατέθηκαν. Και αναφερόμαστε εδώ πέρα απλώς και μόνο σε μία γνωμοδότηση, έτσι μην το ξεχνάμε δεν εξετάζουμε αυτή τη στιγμή κάποια έκθεση. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η νομοθετική δέσμη. Από τις 473 τροπολογίες καταλήξαμε σε 43 συμβαστικές τροπολογίες κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των σκιωδών εισηγητών. Το μεγαλύτερο τμήμα λοιπόν της δουλειάς έχει ήδη γίνει. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων αυτών γίνανε διάφορες απόπειρες προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμβασμούς, πράγμα το οποίο δεν ήταν εύκολο βέβαια, και αυτό διότι υπάρχει μία απόσταση τοποθετήσεων για διάφορα ζητήματα από τη μία πολιτική ομάδα στην άλλη. Κάθε φορά που συζητούσαμε αυτό το σχέδιο πρότασης, αυτό που είχαμε κατά νου είναι ποιος είναι ο απότερος πολιτικός στόχος αυτής της πρότασης οδηγίας σε σχέση με τη θέση του Συμβουλίου τελικά, η οποία έχει ήδη το οποίο έχει ήδη ταχθεί πέρα αυτή τη πρόταση. Στο παρελθόν είδαμε διάφορες αποτυχίες στα πλαίσια της οδηγίας όσον αφορά την άδεια μητρότητος. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι έπρεπε να θέσουμε τώρα φιλόδο, φιλόδοξους στόχους, υπόψη ότι η άδεια πατρότητα εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, αποκλειστικά μάλιστα. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνουν ένα ελάχιστο επίπεδο λύσεων όσον αφορά την άδεια πατρότητας και τη γονική άδεια. Ξέρετε ότι κάθε χώρα έχει τις δικές της διαπραγματευτικές στρατηγικές. Η έκβαση όμως των διαπραγματεύσεων αυτών θα πρέπει πάντα να οδηγεί σε ελάχιστα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Στα πλαίσια της οδηγίας θέλουμε ελάχιστα κοινοτικά πλέον πρότυπα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα της δικής μου της χώρας, της Πολωνίας. Ορισμένες νομοθετικές λύσεις που έχουν βρεθεί στη δική μου τη χώρα είναι πολύ θετικές. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες που μολονότι έχουν θεσπίσει άδεια πατρότητα ή γονική άδεια, η αμοιβή για τις άδειε αυτές είναι πάρα πολύ χαμηλή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ένα ισότιμο επίπεδο φιλοδοξίας όσον αφορά τις άδειε αυτές. Και θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να διασφαλίσουμε ότι ε, θα ισχύει σε όλες τις χώρες ε, η ιδέα αυτή της γονικής άδειας. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να είμαστε αρκετά συγκρατημένοι στις, ε, στην πολιτική μας βούληση, στις πολιτικές μας φιλοδοξίες. Θα πρέπει να κινηθούμε με τρόπο λογικό και στρατηγικό και θα πρέπει να έχουμε κατά νου πάντα τις βασικές αρχές της ισότητας των δύο φύλων. Αυτή είναι, αν θέλετε, η όλη λογική πίσω από αυτή την πρόταση οδηγίας. Η αποψή μου είναι ότι έχουμε εδώ πέρα δύο βασικούς πυλώνες. Η μη μεταβασιμότητα μεταξύ των δύο γονιών όσον αφορά την γονική άδεια. Αυτός είναι ένας βασικός πυλώνας, μια βασική αρχή. Μη μεταβασιμότητα αυτή είναι η πρώτη αρχή και η δεύτερη αρχή είναι ότι η γονική άδεια σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αμείβεται σωστά. Θα πρέπει να αμείβεται παρκώς. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε και περισσότερους πατέρες να υποφελούνται από την άδεια αυτή και να μην μεταβιβάζεται όλη αυτή η γονική άδεια μόνο στι μητέρε. Θέλουμε να υποφεληθούν από την νέα αυτή διάταξη και οι πατέρες και να είναι σε θέση να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά τους. Ξέρετε ότι πολλέ φορέ οι γυναίκε επιβαρύνονται με επαγγελματικέ ευθύνε, αλλά από την άλλη έχουν και πολλέ άλλε ευθύνε φροντίδα για ηλικιωμένου γονεί, για άλλα εξαρτώμενα μέλη τη οικογένεια. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίζεται ο απαραίτητο χρόνο στι γυναίκε αυτέ και απαραίτητε δυνατότητε προκειμένου να μπορούν να συγκεράσουν και να συμφιλιώσουν ιδιωτική και επαγγελματική ζωή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου όσοι κατέθεσαν τροπολογίε. Σίγουρα το όλο πνεύμα συνεργασία ήταν πάρα πολύ επικοδομητικό και ελπίζω ότι ε, θα καταφέρουμε να υποστηρίξουμε όλες αυτές τις ιδέες που εκφράζονται μέσω των τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε κατά την εβδομάδα του Μαΐου στον, στο Στρασβούργο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους λοιπόν τους συναδέλφους και τη Γραμματεία για την υποστήριξή της. Σας ε, ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε τους κοιόδης ε, εισηγητές και θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ε, άποψη της δικής μου πολιτικής ομάδας. Η ομάδα των σοσιαλιστών θεωρεί ότι μια βασική τροπολογία έχει να κάνει με τον ε, συμβιβασμό που θέλουμε να πετύχουμε για την αμοιβή για κάθε μορφή άδειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν οι άδειε αυτέ δεν συνοδεύονται από την κατάλληλη αμοιβή, σαφώ δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσουν την άδεια αυτή οι γονεί. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει η φυστάμενη κατάσταση και γι' αυτό το λόγο η δική μου πολιτική ομάδα προτείνει να υπάρχει μία αμοιβή η οποία να αντιστοιχεί στο 85% του μισθού. Μολονότι το ποσό αυτό είναι υψηλό, δεν θα πρέπει να χάνουμε από το βασικότερο στόχο της οδηγίας αυτής, ότι θα πρέπει δηλαδή τα βασικά καθήκοντα να επιμερίζονται ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας βέβαια και τις δημογραφικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε και η δική μας σκιώδη συγγήτρια, μπορεί τελικά να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό όσον αφορά την ε, αμοιβή για τις άδειε αυτές. Υποβάλαμε επίσης τροπολογίες όσον αφορά και την γονική άδεια. Εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε εδώ πέρα την, το ηλικιακό όριο των 12 ετών που προβλέπεται. Η γονική άδεια θα πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιηθεί από τους δύο γονείς προτού φτάσει το παιδί την ηλικία των 12 ετών. Επίσης η πολιτική μου ομάδα θεωρεί ότι οι εργοδότες θα πρέπει να αιτιολογούν γραπτός οποιαδήποτε άρνηση παροχής της γονικής αυτής άδειας. Επίσης, ο εργοδότης θα μπορεί να αναβάλει, να μεταθέτει χρονικά μία μόνο φορά τη γονική αυτή άδεια. Επίσης, οι εργαζόμενοι θα πρέπει από την άλλη να ενημερώνουν εκ των προτέρων τον εργοδότη προκειμένου αυτός να μπορέσει τελικά να δώσει αυτή την άδεια. Η ομάδα των σοσιαλιστών επίσης θεωρεί ότι θα πρέπει να λάβουμε περισσότερο υπόψη μας τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ξέρετε ότι αναφέρομαι εδώ πέρα σε επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με δύο-τρεις απασχολούμενους το πολύ. Όσον αφορά τώρα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκεί η κατάσταση είναι διαφορετική, καθότι οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να έχουν ε, από 5 έως 250 εργαζόμενους. Θα πρέπει λοιπόν και αυτές οι επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να είναι σε θέση να παρέχουν αυτή τη γονική άδεια. Όσον αφορά τώρα την περίοδο αρχαιότητος, προτού ένας εργαζόμενος έχει πρόσβαση στην γονική αυτή άδεια, η προβλεπόμενη περίοδος του ενός έτους θεωρούμε ότι είναι αρκετά μεγάλη περίοδος γιατί γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τι σημαντικέ εξελίξει που έχουμε στην αγορά εργασία. Έχουμε πάρα πολλού εργαζόμενου που δεν μένουν ένα ολόκληρο έτο σε μια θέση απασχόληση, αλλά αλλάζουν δουλειά πολύ πιο συχνά. Και α μην ξεχνάμε ότι οι νέοι τελικά είναι αυτοί που αποκτούν παιδιά. Επομένω, η περίοδο αυτή του ενό έτου που προβλέπεται δεν θα είναι σε θέση να εφαρμοστεί πάντα. Όσον αφορά τώρα την αρχή της μη μεταβασιμότητος, Θεωρούμε και εμείς ότι θα πρέπει να έχουμε τέσσερις μήνες για τους πατέρες, τέσσερις μήνες για τις μητέρες, όσον αφορά πάντα τη γονική άδεια. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό, όπως ακούσαμε στις 28 Μαΐου θα ψηφίσουμε στα πλαίσια της Επιτροπής μας. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση η τελική τοποθέτηση της δικής μας Επιτροπής να είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη εν και των διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν με τα κράτη-μέλη. Κύριε Πέτρης Βεστέρα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να επαναλάβω πολλά από τα επιχειρήματα που ανέφερε η συνάδελφος από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί πραγματικά ε, προσπαθεί ε, να συστηματικοποιήσει τη δουλειά της. Αξίζει αναγνώριση και η γνωμοδότηση αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, έχει πάρα πολύ μεγάλη ουσία ε, και δείχνεται πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Ε, νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλη συνένεση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά θέματα που αφορούν περισσότερο, όπως είπε και η Πρόεδρος, ε, τις αμοιβέ. Πώς αμείβονται οι γονικές άδειες, οι άδειες πατρότητας και οι άδειες για τη φροντίδα. Θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια αντικειμενικά, 85% ας πούμε ε, αυτό είναι ο στόχος μας, αλλά πάντα σύμφωνα με τα οικονομικά στάνταρ και τα πρότυπα της κάθε χώρας. Ε, αν πληρώνεται σαν την άδεια αν αμείβεται έτσι η άδεια πατρότητα, θα υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορέ. Γιατί από χώρα σε χώρα διαφέρουν τα πράγματα. Θα πρέπει να είναι συγκρίσιμη λοιπόν η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σοβαρή και πλήρη η διαπραγμάτευση που γίνεται για την γνωμοδότηση, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το στόχο της οδηγία αυτής ε, που είναι να αρθούν τα εμπόδια έτσι ώστε η γυναίκα να μπορεί να έχει πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας με πραγματική ισότητα και ισότητα ευκαιριών. Μεταξύ αυτών των εμποδίων φυσικά είναι και το γνωστό ε, θέμα ε, της ε, εργασιακής και της ιδιωτικής ζωής. Από πλευρά των φιλελευθερών, εγώ έχω επιμείνει πάρα πολύ στο ότι χρειάζεται ορισμός για το πλαίσιο διαπραγμάτευσης της οδηγίας αυτής. Θα πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για συμπληρωματικές άδειες ή δευτερεύουσες άδειες ή επικουρικές ας πούμε άδειες ε, και χωρίς να συζητάμε τις, τις άδειες μητρότητας που ήταν επί χρόνια σε ένα σιρτάρι και δεν έχει δοθεί συνέχεια στη σχετική οδηγία. Δεν μπορούμε να συζητάμε την άδεια πατρότητα, την άδεια τη γονική, την άδεια για φροντίδα και άδεια μητρότητα που είναι. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με τα δευτερεύοντα, α πούμε. Χρειάζεται και ε, το πρωταρχικό να λυθεί όλα τα στοιχεία που αφορούν αυτή την πρόσβαση, την ουσιαστική επαναλαμβάνω της γυναίκας στην αγορά εργασίας, ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την ε, άδεια μητρότητας. Αν θέλετε να την ονομάσουμε έτσι, να την πούμε κάπως αλλιώς. Αλλά σήμερα η άδεια μητρότητας με τον τρόπο που ισχύει είναι του 1992. Ε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τελείως ασύμβατα ε, με τις νέες σκέψεις και τους νέους προβληματισμούς. Υποστηρίζουμε λοιπόν την εισηγητρία και σε αυτό και ε, θέλουμε να υπάρξει αυτό το πλαίσιο, το ενοιολογικό να συμπεριλαμβάνεται και η αδιαμητρότητα. Κάτι άλλο που θέλω να θυμίσω είναι ότι είναι φιλόδοξη αυτή εδώ η γνωμοδότηση, γιατί βεβαίως έχει σημασία, αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστική. Φιλοδοξία λοιπόν και ρεαλισμός θα μας επιτρέψουν να προτείνουμε κάτι που θα πιάσει τόπο και θα έχει πραγματικά προστιθέμενη αξία αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Ο, λόγο ο λόγος του κύριο Χρυσόγωνο που αντικαθιστά την κυρία Κούνεμα. Παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω ελληνικά. Ε, εκ μέρους της ε, Κωνσταντίνας Κούνεβα, σκιώδους εισηγήτριας για το φάκελο, επιτρέψτε μου δύο λόγια, ε, επειδή η ίδια λόγω προβλήματος της υγείας της δεν μπορούσε να παραστεί στη συνεδρίαση. Μιλάμε σήμερα για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά κοινωνικά νομοθετήματα αυτής της θητείας, δηλαδή για την πρόταση οδηγίας για την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Ε, για το θέμα αυτό εργάστηκα και εγώ ως σκιώδης συζητητής στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Η πρόταση οδηγίας για την οποία συζητάμε μας ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση αν αναλογιστεί κανείς πως η Επιτροπή είχε δεσμευτεί ήδη από τις αρχές της θητείας της να φέρει μια νέα πρόταση σε αντικατάσταση της οδηγίας μητρότητας. Μια οδηγία που μετράει ήδη 26 χρόνια ζωής. Το Συμβούλιο έδειξε πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον να εξυγχρονίσει τις διατάξεις για τη μητρότητα το 2000. Δεν επιτεύχθηκε τότε συμφωνία και έτσι η πρόταση αναθεώρησης να βάγισε και μέσω της διαδικασίας refit η Κομισιόν την απέσυρε. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια παρόμοια συγκυρία. Και μάλιστα πριν καν να έχουμε την επίσημη θέση του Κοινοβουλίου που συνομοθετεί για το θέμα αυτό. Στο Συμβούλιο μαθαίνουμε πως επιχειρείται να αποδυναμωθεί η πρόταση λέξη προς λέξη. Το Κοινοβούλιο λοιπόν χρειάζεται να εμφανιστεί με μια ισχυρή θέση και να μην επηρεαστεί από τις ειρήνες του Συμβουλίου στο πλαίσιο μιας φαινομενικής σύγκλησης προκειμένου να μην καταπέσει και αυτή η οδηγία όπως έγινε πριν μερικά χρόνια με την πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για την άδεια μητρότητας. Το πρώτο θέμα, το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, είναι ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η οδηγία αναφέρεται ρητά σε εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, αφήνοντας έρμεα εκατομμύρια συμπολίτες μας που είναι ψεύδο αυτοαπασχολούμενοι ε, ή απασχολούμενοι, όπως τους αποκαλούμε στην Ελλάδα, με μπλοκάκι. Η οδηγία οφείλει να καλύψει το κενό που δημιουργείται για αυτήν την μεγάλη κατηγορία εργαζομένων και γι' αυτό κρίνεται απαραίτητη μια αλλαγή στο άρθρο 2. Η πρόταση Κωνσταντίνα Κωνσταντίνας Κούνεβα, η οποία κατατέθηκε με την τροπολογία της 221, καλύπτει πλήρως την ανάγκη αυτή, εισάγοντας μια γλωσσικά ουδέτερη διατύπωση, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί τον ορισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό προσδιορίσε τον εργαζόμενο ή την εργαζόμενη στις υποθέσεις Λόρι Μπλουμ και Γκέντς. Το δεύτερο σημαντικό σημείο το οποίο έχει θίξει η Κωνσταντίνα Κούνεβα με τις τροπολογίες της είναι το επίπεδο αμοιβή της άδειας πατρότητας και της γονικής άδειας. Η πρόταση για αμοιβή στο επίπεδο του επιδόματος ασθενείας είναι προσβλητική τη δεδομένη χρονική στιγμή που η κοινωνική Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση. Πόσο κοινωνικός είναι ο περιβόητος πυλώνας που ευαγγελίζεται η Επιτροπή όταν το πρώτο νομοθέτημα που βλέπει το φως της δημοσιότητας στο πλαίσιο του αντιμετωπίζει τους γονείς που φροντίζουν τα παιδιά τους ως άρρωστους και γι' αυτό τους προτείνει άδεια σε επίπεδο επιδόματος ασθενείας. Οι γονείς που μεγαλώνουν παιδιά δεν είναι άρρωστοι. Είναι εργαζόμενοι που προσδοκούν να αναθρέψουν τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια και αναλόγως αξιοπρεπής να είναι και οι συνθήκες εργασίας τους. Χρειάζεται επομένως καλά αμοιβόμενη άδεια πατρότητας και γονική άδεια αυτή θα πρέπει να είναι η θέση με την οποία θα μετάσχει το Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις. Το τρίτο σημαντικό σημείο στο οποίο χρειάζεται να στραφεί η προσοχή των εισηγητών είναι το ζήτημα της ευελιξίας. Η πρόταση οδηγίας καθιερώνει την ευέλικτη εργασία με έναν τρόπο συγκαλυμμένο, προβάλλοντάς την σαν το μοναδικό εργαλείο για να ισορροπήσουν οι γονείς την προσωπική και επαγγελματική ζωή. Παραπέρα, η οδηγία απορριθμίζει ακόμη περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις μέσα από το άρθρο 9, το οποίο αναφέρεται στο δικαίωμα των γονέων με παιδιά ηλικίας έως 12 ετών να έχουν ευέλικτο ωράριο, χρονοδιάγραμμα ή τόπο εργασίας, όμως ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να εγκρίνει το αίτημά τους. Αυτή την κερκόπορτα της ευελιξίας πρέπει να την κλείσουμε, προβλέποντας ρόλο για τα συνδικάτα και για τις συλλογικές συμβάσεις. Επίση, χρειάζεται να τροποποιηθεί η αναφορά σε αυτήν σε όλο το κείμενο τη πρόταση οδηγία. Δεν θα πρέπει να μιλάμε για ευελιξία, αλλά για προσαρμοζόμενε στον εργαζόμενο ρυθμίσει εργασία. Σχετικέ τροπολογίε έχουν κατατεθεί από την Κωνσταντίνα Κούνεβα. Τέλο, ένα σημαντικό σημείο που η Κωνσταντίνα Κούνεβα έχει αναδείξει μέσω των τροπολογιών τη και χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά είναι η νεοεισαγόμενη άδεια για του φροντιστές στο κείμενο της οδηγίας χρειάζεται να αποσαφινιστεί ο όρος φροντιστής ή φροντίστρια, όπως αυτός ερμηνεύεται με βάση το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η αποσαφήνιση του ορισμού της άδεια φροντίδας είναι απαραίτητη, καθώς είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται σχετικός όρος στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εποφελούμενοι από την άδεια αυτή πρέπει να είναι ξεκάθαρο πως είναι εργαζόμενοι και εργαζόμενες που παρέχουν άτυπα υποστήριξη και φροντίδα στα μέλη της οικογένειάς τους στο πλαίσιο της καλώς νοούμενης οικογενειακής σχέσης. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια ορολογία που θα εισάγει διάκριση μεταξύ των ατόμων που παρέχουν άτυπα φροντίδα εκτός πλαισίου επαγγελματικής, τυπικής ή de facto απασχόλησης σε συγγενείς, παιδιά ή εξαρτώμενα άτομα του οικογενειακού ή διευρυμένου οικογενειακού περιβάλλοντος τους αφενός και αφετέρου σε αυτούς οι οποίοι παρέχουν επαγγελματικά υπηρεσίες φροντίδας. Σε μια χρονική συγκυρία που επιφυλάσσει για τους πολίτες της Ευρώπης πληθώρα υποχρεώσεων, απαιτήσεων, δεσμεύσεων και προκλήσεων, η ισορροπία ανάμεσα στην εργασιακή και την προσωπική ζωή έχει καταστεί κυρίαρχο ζητούμενο και επιτακτική ανάγκη. Και αυτή η πρόταση οδηγίας είναι ευκαιρία προκειμένου να δείξουμε στους πολίτες που μας εξέλεξαν πως η φωνή τους δεν χάθηκε και πως η κοινωνική Ευρώπη δεν συνιστά όραμα, αλλά άμεσα εφαρμοστέα πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Νόχιλα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σκιώδης. Θέλω όμως να επισημάνω ένα σημείο. Μάλλον δεν θα πείσω κανέναν. Παρ' όλα αυτά θέλω να το και αυτό είναι η δυνατότητα μεταβίβασης του χρόνου. Αυτή η δυνατότητα σημαίνει ότι στην πράξη για άλλη μια φορά θα παίρνουν την άδεια την γονική εκείνη που έχουν μικρότερη αμοιβή το ξέρουμε από την εμπειρία μας και στη Γερμανία και επίσης θα σημαίνει ότι οι εργοδότες για άλλη μια φορά θα έχουν, την άποψη ότι αυτή η άδεια θα αφορά κατά κύριο λόγο τις γυναίκες και αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην επαγγελματική τους εξέλιξη και σταδιοδρομία. Γιατί θα σου λέει θα κάνει παιδιά, άρα ε, ε, δεν με συμφέρει. Το δείχνουν και οι στατιστικές αυτό. Σε κάποιες χώρες υπάρχει αυτή η δυνατότητα μεταφοράς της γονικής άδειας και σε, η εμπειρία σε όλες αυτές τις χώρες δείχνει ότι τελικά οι γυναίκες είναι αυτέ που την παίρνουν. Αν όχι στο πρώτο παιδί, τουλάχιστον στο δεύτερο ή στο τρίτο. Ξέρω ότι είναι μειοψηφική η θέση μου. Και το δέχομαι, εντάξει. Αλλά θέλω να το πω. Αν θέλουμε από τη σκοπιά της εξίσωσης των δύο φύλων, μαζί με την κοινωνική πολιτική που θέλουμε να ασκήσουμε, που όλα αυτά σωστά είναι, και δεν θέλω να διαφωνήσω με τίποτα από όλα όσα ακούστηκαν σήμερα. Αλλά αν θέλουμε από άποψη πολιτική για τι γυναίκε, τότε πρέπει να μην υπάρχει δυνατότητα μεταφορά. Όχι για να στραγγαλίσουμε τι γυναίκε, αλλά για να εξασφαλιστεί η ίση θέση των γυναικών και των ανδρών. Που να σημαίνει για τον εργοδότη ότι το να προσλάβω έναν άνδρα σε υψηλή θέση ενέχει τον ίδιο κίνδυνο να μου φύγει σε γονική άδεια όπω αν, πάρω, αν προσλάβω γυναίκα. Αυτό ήθελα απλά να το ξαναθέσω εδώ στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την συζήτηση που γίνεται σήμερα και για τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει πολλοί ευρωβουλευτές στο θέμα αυτό. Θέλω να τονίσω ένα θέμα μόνο, γιατί υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Θέλω να πω λοιπόν ότι η πρόταση αυτή πραγματικά μπορεί να αποδείξει στους πολίτες της Ένωσης τι ακριβώς σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο κοινωνικό μέτωπο. Η ισορροπία ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής είναι θέμα που ε, απασχολεί ε, πάρα πολλού ανθρώπου. Αν σήμερα βρεθήκατε στο αεροδρόμιο των Βρεξελών, θα είδατε ότι υπάρχει μια απεργία που, έχει ω θέμα τη ακριβώ αυτό. Τα δικαιώματα λοιπόν που θεσπίζει αυτή η οδηγία θα έχουν ε, θετικέ επιπτώσει στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων και γι' αυτό και είμαστε ευγνώμονε ε, προ την εισηγήτρια για το γεγονό ότι διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος των φιλοδοξιών ε, που είχαμε και εμείς είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο και για τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν με το Συμβούλιο. Γι' αυτό και θέλω να κάνω αυτή την έκκληση προς εσάς να διατηρήσουμε το επίπεδο ε, φιλοδοξίας, ταυτόχρονα όμως παραμένοντας ρεαλιστές, όπως είπαν και κάποιοι από τους κοιόδησίτες, ε, ε, να αποφύγουμε αυτό που συνέβη με την οδηγία για την ε, άδεια μητρότητα. Πρέπει λοιπόν δηλαδή πραγματικά να παραμείνουμε ρεαλιστέ. Από πλευρά κομισιών αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είμαστε στη διάθεσή αν θέλετε να συζητήσουμε, να διευκρινίσουμε θέματα, να δούμε συμβαστικέ διατυπώσει αν το επιθυμείτε. Είμαστε στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην κυρία Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω από το τελευταίο σχόλιο που έκανε η κυρία Νόιχλ. Ίσως υπήρξε κάποια ε, παρανόηση στην ε, ε, συζήτηση. Η μη δυνατότητα μεταφοράς των ε, γονικών αδειών, η ξεχωριστή άδεια για τον πατέρα και την μητέρα είναι η βασική αρχή. Και υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία ε, υπέρ της μη μεταβιβασιμότητας διότι η δυνατότητα μεταφοράς θα σήμαινε ότι στην πραγματικότητα θα κατέλεγαν οι γυναίκες να τη χρησιμοποιούν την άδεια αυτή. Στην Πολωνία υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς και είναι σαφές σε όλους ότι ε, κατά κύριο λόγο και στη μεγάλη τους πλειοψηφία γυναίκες είναι αυτές που ε, χρησιμοποιούν την άδεια αυτή. Τώρα, προφανώς κάποιος πρέπει να φροντίσει το παιδί αφού γεννηθεί. Και αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Ωστόσο, συνήθως το βάρος αυτό πέφτει στους ώμους των γυναικών. Και οι εργοδότες, για τους εργοδότες μάλλον, οι γυναίκες αποτελούν ρίσκο, κίνδυνο, γιατί μπορεί να σου πάρει άδεια μητρότητα, αν την προσλάβεις. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε σε αυτό που είπατε κι εσείς, τη μη μεταβιβασιμότητα των αδειών. Αναδρομικά λοιπόν και έχοντας κατά νου και τις συζητήσει που είχαμε με τους σκιώδεις, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της απαγόρευσης μεταφοράς των αδειών από τη μητέρα στον πατέρα και αντίστροφα. Και υπέρ της διακριτότητας των δύο αδειών. Τώρα, να περάσω και σε κάποια άλλα θέματα. Κυρία Πρόεδρε, εσείς αναφερθήκατε σε ορισμένα σημεία που σχετίζονται με την ανάγκη ε, που πόσο χρειάζεται κανείς να έχει δουλέψει για να μπορεί να πάρει μια άδεια ε, Εδώ εμείς αναφέρουμε ε, ένα χρόνο. Αυτό όμως δεν είναι ακριβές, γιατί η πρόταση προτείνει ως maximum τον ένα χρόνο. Τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα από εκεί και πέρα να θεσπίσουν και μικρότερους χρόνους. Η πρόταση λοιπόν αναφέρεται στο ότι οι αποφάσεις των κρατών μελών δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε κάποιες χώρες λοιπόν ε, υπάρχουν ε, δυσμενέστερες ε, συνθήκες για να πάρει κανείς την άδεια ε, μητρότητας. Φανταστείτε δηλαδή ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δεν θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν ε, τις δυνατότητες που τους δίνει η οδηγία. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να επιμείνουμε στον ένα χρόνο, αλλά ως μέγιστο όριο που μπορεί να θεσπιστεί για να μπορεί κανείς να θεμελιώσει δικαίωμα λήψης άδεια μητρότητα. Επίσης, συμφωνώ με την Πρόεδρο ότι η μη μεταβιβασιμότητα και το γεγονός ότι πρόκειται για αμοιβόμενη άδεια είναι δύο στοιχεία που πρέπει ε, να εξασφαλιστούν απολύτως. Υπάρχει όμως μια μικρή απόκληση θέσεων Ω προ το επίπεδο της αμοιβή. 70% είπε το ΕΛΚ, 60% έχουν προτείνει άλλε ομάδες, κάποια ομάδα πρότεινε 85%. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό και ω προ το ποσοστό. Εγώ θα προτιμούσα βεβαίω να κινηθούμε πιο, πολύ, πιο κοντά στο 70%. Το 85% δεν μου φαίνεται ρεαλιστικό. Πάντω υπάρχει συμφωνία από ό,τι φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει το σημείο αναφοράς που προτείνει η Κομισιόν. Γιατί η Κομισιόν ε, προτείνει την άδεια ε, ασθενείας ως σημείο αναφοράς για να υπολογίζεται η άδεια μητρότητας. Εμείς ως Επιτροπή Γυναικών θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό και να λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός μισθός, η πραγματική αμοιβή που παίρνει η εργαζόμενη ή ο εργαζόμενος. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικότερο και πολύ καλύτερο. Γιατί κάποιες φορές η άδεια ασθενεία ε, αντιστοιχεί μόλις το 40% του μισθού που παίρνεις στη δουλειά σου. Άρα για μας είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει και αυτό, το σημείο αναφοράς, το, η βάση ε, η οποία θα χρησιμοποιείται για να υπολογίζεται η αμοιβή που θα λαμβάνει μια γυναίκα ή ένας άνδρας κατά την γονική άδειά του. Επίσης, Συμφωνώ με την... Με τα όσα ακούστηκαν σχετικά με την, την ε, ανάγκη να υπάρχει υποχρέωση εργοδότης να απαντά γραπτός σε περίπτωση που αρνείται να παράσχει σε εργαζόμενο του άδεια πατρότητας ή μητρότητας. Αυτή, ε, αυτή η μητροτητας αυτη είναι πολύ, ε, η διάσταση είναι πολύ σημαντικό, σημαντική Βεβαίω, για τους εργαζόμενους. Πρέπει όμως να οριστεί και ένας ανώτατος αριθμός ε, φορών που θα πρέπει ένας εργοδότης να προβαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ξέρετε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν και κάποιες, κάποιες, κάποιους περιορισμούς αντικειμενικούς ως προς τις δυνατότητες τους να ε, προβαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία. Ελάχιστα λοιπόν να είναι τα, τα πρότυπα που θεσπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από εκεί πέρα τα κράτη-μέλη να είναι ελεύθερα βεβαίως να θεσπίζουν και αυστηρότερες ε, διαδικασίες προκειμένου να προστατεύονται και οι εργαζόμενοι αλλά και οι επιχειρηματίες έχοντας κατά νου πάντοτε ιδίως τις πολύ πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις δυνατότητες ή τον περιορισμό των δυνατοτήτων τους. Όσον αφορά την πρόταση της ΓΚΟΕ ε, εγώ βεβαίως δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας γιατί θεωρώ ότι ε, ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας θα μας οδηγήσει αναγκαστικά σε ε, αποτυχία όπω συνέβη και με την οδηγία για την άδεια μητρότητα. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξη, Σημείο 7 Προπολογισμό 2019, εντολή για τον τριμερή διάλογο. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μπιόρκ, την εισηγήτριά μα. Ε... Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε η δυνατότητα να σας παρουσιάσω αυτό το κείμενο εξ τη της Επιτροπής Γυναικών. Είναι σημαντικό και η Επιτροπή Γυναικών να συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή και στη συζήτηση για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και για τον προπολογισμό του 2019. Ψηφίσαμε άλλωστε και για τα πιλωτικά προγράμματα και αυτό το αναφέρω στο σχέδιο της γνωμοδότησής μου. Είναι σύντομη γνωμοδότηση. Τρία πράγματα είναι για μένα σημαντικά. Το gender mainstreaming, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές. Αυτό θα πρέπει να είναι ε, μια κεντρική ιδέα σε όλο τον προπολογισμό και να αποκτήσει και πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα. Και όλα αυτά θα πρέπει να παίξουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο στο μέλλον και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ένα άλλο κομβικό σημείο κατά την άποψή μου είναι θα πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο ε, στο κράτος πρόνοιας, στη φροντίδα, ε, στην εκπαίδευση ε, για επαγγελματά υγείας και φροντίδας χρειάζεται μεγαλύτερη πρικοδότηση εκεί από τον προϋπολογισμό. Και επίσης πιστεύω ότι να ενισχύσουμε το ρόλο και τη θέση των γυναικών, ε, η προστασία της υγείας και των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων με αντίστοιχη χρηματοδότηση. Γιατί και εκεί χωλένει ο προϋπολογισμός και θα πρέπει να φροντίσουμε τα ελλείμματα αυτά να καλυφθούν. Κατά τα άλλα, εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε το Ινστιτούτο Φίλου που είναι ένα παρατήριο της κατάστασης ε, που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, συγκεντρώνει στατιστικά και αριθμητικά στοιχεία. Θα κάνω και τροπολογίες εγώ ε, για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και επίσης ε, για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών ε, στα διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι βλέπουμε ότι το περιθώριο ελιγμών και για τις γυναίκες περιορίζεται συνέχεια. Και θα καταθέσουμε και εκεί τροπολογία σχετική ε, για την έμφυλη βία. Μέχρι τώρα νομίζω δεν το έχουμε δει στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. η βία κατά των γυναικών πραγματικά έχει να κάνει με το φίλο τους, με κάποιες τρευλές αντιλήψεις, προκαταλήψεις, παραδόσεις κτλ. Αυτά. Περιμένω και τις δικές σας τροπολογίες και ελπίζω να ενισχύσουν την ε, γνωμοδότησή μας. Σκιώδεις συζήτητες, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Πίνα Πιτσέρνο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο κυρία Μπιόρκ για την εξαιρετική της εργασία. Θεωρώ πραγματικά ότι έχει επικεντρωθεί σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία των γυναικών. Σίγουρα το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ζήτημα μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές και στα πλαίσια της Επιτροπής μας. Παρ' όλα αυτά, είναι μόνο μία πτυχή αυτή τις εργασίες που θα πρέπει να κάνουμε για τον κοινοτικό προπολογισμό σε σχέση με τις γυναίκες. Το έχω ξαναπεί αυτό και στο παρελθόν, όταν για πρώτη φορά συζητήσαμε τους στόχους του προπολογισμού για το 2019 στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που κάναμε στις 25 Απριλίου. Θα θυμάστε ότι τότε είχα πει ότι ο ρόλος και η χειραφέτηση των γυναικών θα πρέπει να μπορεί να προωθηθεί και μέσω της οικονομικής χειραφέτησής τους. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πόρους οικονομικούς για να αυξήσουμε την απασχολησιμότητα των γυναικών ζήτημα το οποίο μας έχει απασχολήσει επανειλημμένο στα πλαίσια της Επιτροπής μας και ζήτημα το οποίο εγώ δεν θα σταματήσω να προωθώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η απασχόληση των γυναικών οδηγεί τελικά στην ίδια την αυτονόμηση, την ανεξαρτησία και την χειραφέτηση των γυναικών. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν οι γυναίκες να λειτουργήσουν αυτόνομα και ανεξάρτητα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το στόχο αυτό. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε όλο το ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με τη μετανάστευση. Ξέρετε ότι ε, ακόμα και η ασφάλεια και η αναπτυξιακή βοήθεια που έχει να κάνει με τη μετανάστευση έχει μια διάσταση φύλου που είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει δηλαδή να καταφέρουμε να προβλέψουμε συγκεκριμένη υγειονομική υποστήριξη για τις γυναίκες μετανάστες συγκεκριμένη υποστήριξη οικονομική για την ενσωμάτωσή τους, για την κατάρτισή τους. Εγώ επίσης, και το ξαναλέω σήμερα, θα ήθελα να έχουμε και τα απαραίτητα κονδύλια προκειμένου το πρόγραμμα Δάφνη το οποίο είδαμε από το 2000 μέχρι το 2014 να μπορούμε ουσιαστικά να το ενεργοποιήσουμε και για το μέλλον, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το σημαντικότατο έργο του προγράμματος αυτού προκειμένου να καταφέρουμε να προστατεύσουμε περισσότερο τις γυναίκες από φαινόμενα όπως εμπορία ανθρώπων ή σεξουαλική κακοποίηση. Θέλω μη τι άλλο να καταφέρουμε να αναστήσουμε κάπως το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα Δάφνη. Όλα τα στοιχεία αυτά θα μπορέσετε να τα δείτε στα πλαίσια των τροπολογιών που θα καταθέσω και προσβλέπω σε μια επικοτομητική συνεργασία με την εισηγήτρια. Σας ευχαριστούμε κύριε Πιτσέρνο, λέει πρόεδρος. Δεν έχουμε άλλους ομιλητές. Σας υπενθυμίζω ότι 18 Μαΐ 12 το μεσημέρι είναι καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών. Στις 10 η ώρα προβλέπεται τώρα η συνεδρίαση των συντονιστών. Σε λίγα λεπτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ.